Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, με μεγάλη μου τιμή δέχομαι εδώ τον Dr. Ντένις Δημουτβέγκε, Μαντελέν Καμπέμπο Καμπόι, από τη, δημοκρατική, από τη Δημοκρατία του Κονγκό. Τους καλωσορίζω εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Cher Καλώς ορίσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και να πιστέψτε με, κύριε δόκτωρα Μουκβέγγε, προτού τιμήσω την ε, συνεισφορά σας. Επιτρέψτε μου να τιμήσω και κάποιους άλλους προσκεκλημένους που ε, διακρίθηκαν για την ελευθερία σκέψης τους, μεταξύ αυτών και οι εκπρόσωποι εκπρόσωπος πρόσωπος ε, Ελγζαμπέτα εκπρόσωπο της Επανάστασης ε, στο Μαϊντάν από την Ουκρανία. Σας καλωσορίζω εκ βάθους καρδίας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εσείς κυρία Σερπετενικόβα και οι συνάδελφοί σας, οι φίλοι και οι φίλοι σας έδεξτε ε, τεράστιο θάρρος και τόλμη και με κίνδυνο τη ζωή σας ε, αγωνιστήκατε για το μέλλον της χώρας σας. Βγήκατε στους δρόμους για μια δημοκρατική και ελεύθερη Ουκρανία και γι' αυτό λοιπόν σας ε, επιδεικνύουμε την πλήρη υποστήριξή μας και αλληλεγγύη μας. Καλώς ορίσατε. Να καλωσορίσω και την Άρα Γιούρους, ε, κυρία Γιούνους. Ήρθατε εδώ στο Στρασβούργο για να εκπροσωπήσετε τη μητέρα σας, αλλά είναι Γιούνος, η οποία δεν μπορεί να είναι μαζί μας, γιατί ακόμα είναι υποκράτηση σας. Καλώς ορίζω, αγαπητή κυρία Γιούνος. Η κυρία Γιούνος εδώ στο Κοινοβούλιο ε, προτάθηκε για το βραβείο Ζαχάροφ ως ιδρύτρια του θεσμικού οργάνου για την ελευθερία και τη δημοκρατία, για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Αζερμπαϊτζάν, τα οποία και προασπίστηκε με θάρρος και με τόλμη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καλέ την κυβέρνηση στο Αζερμπαϊτζάν αυτή την αθώα γυναίκα της οποίας η υγεία έχει επιδεινωθεί δραματικά να την απελευθερώσει άμεσα και θα ήθελα εδώ να προσθέσω το εξής. Προσπαθήσαμε να αποστείλουμε στο Αζερβαϊτζάν ε, κοινοβουλευτική αποστολή για να επισκεφτεί την κυρία Γιούνος. Μέχρι σήμερα δεν το πετύχαμε, γι' αυτό λοιπόν ρητά διαμαρτύρομαι εδώ. Οι συνάδελφοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην κυρία Γιούνος και καταγγέλλω το γεγονός ότι δεν το έχουν λάβει αυτή την πρόσβαση έως τώρα. Αυτό δεν είναι αποδεκτό. Και γι' αυτό το γεγονός ότι είναι εδώ η κόρη σας σήμερα αποτελεί ένα σύμβολο. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, πολύ καλύτερα από ότι θα μπορούσα εγώ να σας περιγράψω την εργασία του κυρίου Μουκβέγκε, θα σας το περιγράψει ένα σύντομο φιλμ, το οποίο θα ήθελα να σας δείξω πρωτού συνεχίσω. Uh, Οι εντυπωσιακέ αυτές εικόνες που μας ταράζουν λένε πολλά για σας ε, κύριε δόκτωρα Μουκβέγκε. Ένας ε, συναρπαστικός άνθρωπος ο οποίος έχει αφαιρέσει τη ζωή του για τον αγώνα προς τη δικαιοσύνη. Ένας ε, γιατρός ο οποίος ακούραστα φροντίζει τους ασθενούς του και στις χειρότερες δυνατές συνθήκες προσπαθεί να απαλύνει τον τεράστιο πόνο τους και παρόλα αυτά δεν μπορούμε καν να φανταστούμε την εξαθλίωση την οποία βλέπετε κάθε μέρα στη δουλειά σας στο νοσοκομείο που έχετε ιδρύσει με τα χέρια σας εξ ονόματος των συναδέλφων μου σας εκφράζω τον θαυμασμό και τον βαθύ σεβασμό προς το πρόσωπό σας για αυτά που κάνετε κάθε μέρα αντί να αποτάσσεστε όλα αυτά τα πράγματα και να γυρνάτε το βλέμμα σας έχετε διαμορφώσει το έργο σας ως ένας ακούραστος υπέρμαχος για τις γυναίκες, για τα κορίτσια εκείνα τα οποία είναι θύματα σεξουαλικής βίας. Το πόνο αυτών των γυναικών, αμέτρητων γυναικών και κοριτσιών τον έχετε απαλύνει. Τους έχετε την βοηθείας για τα τραυματισμένα σώματά τους, για τις τραυματισμένες ψυχές τους. Ακούραστα Συνεχίζεται να καταγγέλλεται τη σεξουαλική βία ως όπλο του πολέμου κατά των αθώων και ότι αυτές οι ακλειότητες αποτελούν όχι μόνο μονομένα περιστατικά, αλλά τμήμα μια στρατηγική. Οι βιασμοί πάντα είναι απάνθρωποι και βίαιοι, τις τους καταδικάζουμε, αλλά θα πρέπει τα λόγια αυτά να τα ακολουθήσουν και πράξεις. Αυτό κυρίες και κύριοι σημαίνει ότι αυτή η ατιμορρησία η οποία de facto ισχύει σε περιπτώσεις ένοπλων σειράξεων θα πρέπει να λάβει επιτέλους τέλος. Όταν ε, οι βιασμοί διατάσσονται από τους ε, ανώτερους, πρόκειται για έγκλημα πολέμου και τότε τα εγκλήματα πολέμου θα πρέπει να τιμωρούνται ως τέτοια, ως εγκλήματα πολέμου. Και ακόμη στην ε, δημοκρατία του Κονγκού, του Κονγκό γίνεται μαζική βιασμοί. Αναρρύθμιτες γυναίκες έζησαν τα ίδια πράγματα στη Συρία, στο Ιράκ, στην Ρουάντα, στην Βοσνία, Ζεγοβίνη και σε άλλες περιοχές εμπόλεμων σειράξεων. Και σχεδόν όλα αυτά τα εγκλήματα έμειναν ατιμόρυτα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την κυβέρνηση του Κονγκό όπως και τις κυβερνήσεις των άλλων χωρών να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους προκειμένου να σταματήσουν άμεσα οι βιασμοί για να σταματήσει αυτή η ατιμορρησία για τους βιαστές και να κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου οι γυναίκες να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο δικαστικό σύστημα. Αξιότιμε δόκτωρα Μουκβέγγε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το βραβείο Σαχάροφ τιμά την ελευθερία σκέψεως και τιμά την αξιοθαύμαστη εργασία σας ως ε, γιατρός και ως υπέρμαχος της αξιοπρέπειας της, ε, των γυναικών για την ισότητα και την δικαιοσύνη στη χώρα σας. Ελπίζω από κοινού να καταφέρουμε να ευαισθητοποιήσουμε παραπάνω τον κόσμο σε ό,τι αφορά τη χρήση βιασμών ως όπλο πολέμου. Ένα φρικιαστικό έγκλημα το οποίο με όλες τις δυνάμεις μας από κοινού πρέπει να καταπολεμήσουμε για να το εκριζώσουμε. Χθε. Δόκτωρα Μουκβέγκε, είπατε μια πρόταση εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η οποία με εντυπωσίασε ιδιαίτερως. Παραθέτω. Ότι αναγνωρίζετε όλες αυτές τις γυναίκες, όλα αυτά τα κορίτσια Στη χώρα σας, σε όλες τις χώρες του κόσμου, τους αναγνωρίζετε λοιπόν το καθεστώς του θύματος και οφείλουμε να αποδώσουμε δικαιοσύνη. Είμαι περήφανος λοιπόν κύριε και κύριοι για το γεγονός ότι φέτος αποδίδουμε Απονέμουμε το, το βραβείο Ζαχάροφ στον δόκτωρα Μουκβέγγε από το Κονγκό. Κύριε ε, αξιότιμε δόκτωρα Μουκβέγγε, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αξιότιμοι προσκεκλημένοι. Με πολύ μεγάλη ταπεινότητα και με μεγάλη ελπίδα λαμβάνω σήμερα το διακεκριμένο βραβείο Ζαχάροφ για την ελευθερία του πνεύματος. Φέτος, Είχατε την εκατοστή, ε, συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από την ε, έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Ευρώπη νόμιζε τότε ότι θα ήταν ο τελευταίος πόλεμος και ότι ο πολιτισμός θα θριάμβευε. Δυστυχώς, όπως είδαμε, 30 χρόνια αργότερα η ανθρώπινη τρέλα πάλι κατέλησε τον πλανήτη μας. Έκτοτε όμως με το πέρας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου έχετε κάνει την επιλογή ε, να κινηθείτε προς την ειρήνη, να ζήσετε μαζί, όλοι μαζί σε μια κοινωνία η οποία θα προσανατολιζόταν προς την ελευθερία και την ευημερία στο σημερινό πλαίσιο ασφάλεια, το οποίο είναι όλο και πιο ασταθέ, όπου οι αιστείες κρίση πολλαπλασιάζονται και κυρίω στις περιοχέ που γυτνιάζουν άμεσα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ήθελα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο να ευχαριστήσω θερμά τους εκλεγμένους αντιπροσώπους των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι ε, κατάφεραν να διαφωτίσουν, να ρίξουν φως στην ανθρώπινη τραγωδία την οποία βιώνουν οι γυναίκες που είναι θύματα βιασμών και σεξουαλικής βίας ε, στην, ε, στα ανατολικά της Δημοκρατίας του Κονγκό. Σε έναν κόσμο όπου έχουν αντιστραφεί οι αξίες, όπου η βία είναι καθημερινότητα και μάλιστα παίρνει μορφές αποτρόπες, το να αρνείται κανείς τη βία, αυτό σημαίνει ότι είναι αντιφρονών. Εφιστώντας την προσοχή ολόκληρου του κόσμου στην ανάγκη να προστατευτούν οι γυναίκες σε περιόδους ενόπλων συγκρούσεων, εσείς κάνοντας αυτό αρνηθήκατε το προσωπείο της αδιαφορίας έναντι ε, μίας από τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές καταστροφές της σύγχρονης εποχής. Επιβεβαιώσατε και υπογραμμίσατε ότι η επίλυση των συγκρούσεων στην περιοχή των μεγάλων λιμνών και η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η προώθηση των δημοκρατικών αρχών ήταν, είναι και θα παραμείνουν προτεραιότητα για την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική. Με αυτό το βραβείο αποφασίσατε να καταστήσετε πολύ πιο ορατό ε, τον αγώνα που κάνουν οι γυναίκες στο Κονγκό εδώ και 15 χρόνια ώστε να αναγνωριστεί η οδύνη που βιώνουν, η αξιοπρέπεια και το θάρρος ε, που μαρτυρούν. Κύριε Πρόεδρε, η περιοχή όπου ζω είναι μία από τις πιο πλούσιες στον πλανήτη μας. Ωστόσο, η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων στην περιοχή αυτή διαβιεί σε καταστάσεις ακραίας φτώχειας λόγω της ανασφάλειας και της κακής διακυβέρνησης. Το σώμα της γυναίκας έχει καταστεί πραγματικό πεδίο μάχης και ο βιασμός χρησιμοποιείται ως όπλο πολέμου. Αυτό έχει πολλαπλές συνέπειες με πολύ μεγάλο αντίκτυπο στο σύνολο της κοινωνίας. Έχει διαραγεί ο οικογενειακός ιστός, όπως επίσης και ο κοινωνικός ιστός. Οι ολόκληροι πληθυσμοί έχουν ε, υποβληθεί σε καθεστώς δουλείας και έχουν αναγκαστεί, να εξοριστούν. Μέσα σε μια οικονομία η οποία είναι ιδιαίτερο στρατικοποιημένη, όπου ο νόμος των ε, πολέμαρχων είναι αυτός που συνεχίζει να εφαρμόζεται από τη στιγμή που απουσιάζει το κράτος δικαίου. Είναι μια στρατηγική πολέμου η οποία είναι δυστυχώς πολύ αποτελεσματική. Οι αρχές του κράτους του Κονγκό και οι θεσμοί, τα θεσμικά όργανα είναι πάρα πολύ ασταθή, πάρα πολύ εύθραυστα ε, στοιχεία του πολιτεύματο και δεν είναι σε θέση να προστατεύσουν τον πληθυσμό ούτε να ικανοποιήσουν τι βασικέ ανάγκε. Κύριε Πρόεδρε, σπάνιε είναι οι μέρε όπου δεν υπάρχει ανθρώπινο δράμα να σημειώνεται στην περιοχή όπου ζω. Για παράδειγμα, την περασμένη εβδομάδα άνω των 50 ατόμων σφαγιάστηκαν με τη ματσέτα στην, επικράτεια του Μπενή στο βόρειο Κίβου. Ε, ξεκυλιάστηκαν έγκυε γυναίκε, ακροτηριάστηκαν μωρά, βρέφη μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 1,5 μήνα 200 άνθρωποι βρήκαν φρικτό θάνατο. Ως ανθρώπινο όν λοιπόν, ως άνθρωπος και εγώ μεταξύ σας θα ήθελα... να έρθει μια μέρα όπου να μην χρειάζεται και να μην υπάρχει λόγος να αναφέρομαι σε τέτοιου είδους φρικτά εγκλήματα με θύματα ε, συμπολίτε μου και συνανθρώπους μου. Πώς μπορώ όμως να σοπάσω ε, όταν εδώ και 15 χρόνια ε, βλέπουμε φρικαλαιότητες τις οποίες ούτε καν το μάτι του χειρουργού δεν μπορεί να συνηθίσει. Πώς μπορώ να σοπάσω όταν οι οικονομικοί λόγοι είναι αυτοί που οδηγούν ε, ε, τους ανθρώπους να προσφύγουν στο βιασμό ως στρατηγική πολέμου. Πώς μπορώ να σοπάσω όταν γνωρίζουμε ότι οι εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας ε, σχεδιάζονται με κίνητρο αμυγός οικονομικό. Κάθε ε, γυναίκα που έχει βιαστεί την ταυτίζω με τη δική μου σύζυγο. Κάθε μητέρα που έχει υποστεί βιασμό την ταυτίζω με τη δική μου μητέρα και κάθε παιδί που έχει υποστεί βιασμό το ταυτίζω με τα δικά μου παιδιά. Πώς μπορούμε άραγε να σοπάσουμε. Ποιος άνθρωπος με συνείδηση θα μπορούσε να σοπάσει όταν του φέρνουν ένα μωρό έξι μηνών με εδίο κατεστραμμένο είτε λόγω βίαιης διείσδησης, ε, είτε λόγω ε, βίαιης χρήσης εχμηρών αντικειμένων είτε λόγω βίαιης εφαρμογής χημικών προϊόντων στην περιοχή. Ήδη μία περίπτωση βιασμού είναι κάτι το πολύ σοβαρό και χρειάζεται δράση από όλους μας. Στη δική μου χώρα εκατοντάδες χιλιάδες γυναίκες έχουν υποστεί βιασμό και χιλιάδες παιδιά έχουν γεννηθεί μετά από πράξη βιασμού. Και μάλιστα εκατομμύρια άνθρωποι έχουν βρει το θάνατο λόγω των ένοπλων συγκρούσεων. Στον υπόλοιπο κόσμο όλοι θα είχαν εκφράσει τον αποτροπιασμό τους. Στη κοινωνία του Κονγκό, όπου λείπουν τα σημεία αναφοράς, οι φρικαλαιότητες οι μαζικές αποτελούν μέρος της καθημερινότητας, αποτελούν μέρος της επικαιρότητα, όσο σαν επρόκειτο καθημερινές ειδήσει που μεταδίδονται, κάτι το οποίο δυστυχώς ε, δείχνει το βαθύ τραύμα που βιώνει αυτή η κοινωνία, που της έχει προκληθεί από την ε, υπερβολική βία από την απουσία πολιτικής ευθύνης και από την άρνηση ε, της ανθρώπινης υπόστασης που μας χαρακτηρίζει, που μας χαρακτηρίζει όλους. Κύριε Πρόεδρε, έχει έρθει πλέον η ώρα να ασχοληθούμε με τις αιτίε. Έχουμε σπαταλήσει πάρα πολύ χρόνο και πάρα πολύ ενέργεια προσπαθώντας να αποκαταστήσουμε τις συνέπειες της, βίας. της βίας. Πρέπει όμως να ασχοληθούμε με τις αιτίε και οι χιλιάδες μαρτυρίες των θυμάτων δείχνουν ότι ο λαός του Κονγκό διψά για δικαιοσύνη, για ειρήνη και φιλοδοξεί να επέλθει επιτέλους η αλλαγή. Υπάρχουν λύσεις και χρειάζονται ε, πραγματική πολιτική βούληση. Είμαστε σε κρίσιμο χρονικό σημείο. Η Συμφωνία Πλαίσιο για την Ειρήνη, την Ασφάλεια και τη συνεργασία που υπογράφει στην Αντίσα Μπέμπα το 2013 δεν πρέπει να παραμείνει ένα απλό ε, φύλλο χαρτί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ιστορικός εταίρος, είναι ο πρώτος συμβάλλον σε επίπεδο βοήθειας. Καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη να δώσουν νέα πνοή στην εφαρμογή αυτής της ε, συμφωνίας ελπίδας. Καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα, να ασκήσει αν θέλετε πίεση σε όλους τους μοχλου οικονομικούς, χρηματοπιστωτικούς, πολιτικού πολιτικούς διπλωματικούς για να συμβάλλει σε μια οριστική λύση της ένοπλης σύγκρουσης στην περιοχή των μεγάλων λιμνών. Στη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό η ενίσχυση του κράτους και η αποκατάσταση της ασφάλειας στα ανατολικά της χώρας αποτελούν υπέρτατη και μεγίστη προτεραιότητα. Η μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας είναι η πιο σημαντική θεσμική μεταρρύθμιση στο επίκεντρο των προσπαθειών που καταβάλλονται ε, έτσι ώστε το κράτος ε, του Κονγκό οι αρχές να καταφέρουν να προστατεύσουν τον άμαχο πληθυσμό, τους πολίτες. Η δικαιοσύνη θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο της ειρηνευτικής διαδικασίας και η καταπολέμηση της ατιμορρησίας για τα τόσο σοβαρά εγκλήματα και μάλιστα τα εγκλήματα που περιέχουν σεξουαλική βία θα πρέπει να είναι ε, ο βασικός μας αγώνας. Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη ούτε οικονομική ανάπτυξη ούτε κοινωνική ανάπτυξη χωρίς σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη χωρίς αποκατάσταση των ε, όσων έχουν επιζήσει από πράξεις βιασμού, χωρίς αποκατάσταση και αποζημίωση των θυμάτων, χωρίς κάθαρση στο δημόσιο τομέα και μάλιστα κάθαρση και προσεκτική εξέταση ε, των δυνάμεων ασφαλείας, χωρίς μηχανισμούς αποκατάστασης της αληθείας έτσι ώστε να ενισχυθεί επιτέλους η εθνική συμφιλίωση. Κύριε Πρόεδρε, τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν μία από τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αποτελούν συνάμα και έναν από τους στόχους που εμπνέουν τις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η προώθηση της ειρήνης, η προώθηση της ανάπτυξης, η ενίσχυση των δημοκρατικών αρχών και των, του κράτους δικαίου. Ε, φρονώ ε, με κάθε ταπεινότητα ότι, με κάθε ταπεινότητα, με συγχωρείτε, ότι αυτή είναι η πραγματική προστιθέμενη αξία που κομίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τους υπολείπους διεθνείς εταίρους. Η Realpolitik δείχνει πολύ συχνά ότι ε, τα γεωστρατηγικά και οικονομικά συμφέροντα παίρνουν το προβάδισμα έναντι του σεβασμού και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δυστυχώς. Το σχέδιο κανονισμού ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι όπως ε, προβάλλεται και παρουσιάζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για υπεύθυνη προμήθευση σε ορυκτό πλούτο είναι ένα σχέδιο κανονισμού που θα εξετάσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει λοιπόν κατά τη γνώμη μου να περιλαμβάνει μια δεσμευτική διάσταση και να στοχεύει και τα έτοιμα τελικά προϊόντα στη Δύση καθώς και τις βασικές πρώτες ύλες στην Αφρική. Εκφράζω την επιθυμία ο καθένας από εμάς να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να υπάρχει συνοχή μεταξύ των οικονομικών πολιτικών από τη μία και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την άλλη. Έτσι ώστε η ανθρώπινη αξιοπρέπεια να βρεθεί επιτέλους στο επίκεντρο των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών ε, φιλοδοξιών. Η χώρα μας έχει πάρα πολύ μεγάλο δυναμικό. Με ένα πιο υπεύθυνο και πιο διαφανές εμπόριο, αν θέλετε, το Κονγκό μπορεί, έχει ενδογενείς δυνατότητες για ανάπτυξη, χάρη στους πολύ πλούσιους φυσικούς του πόρους και χάρη επίσης και στους ανθρώπινους πόρους του, που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν σήμερα, στο πλαίσιο ε, το, που, στο, σε ένα πλαίσιο κατά το οποίο δεν έχουμε ούτε πόλεμο αλλά ούτε και ειρήνη. Κύριε Πρόεδρε, το βραβείο που μου δίδεται δεν θα έχει καμία σημασία για τις γυναίκες που είναι θύματα σεξουαλικής βίας παρά μόνο εάν μας συνοδεύσετε σε αυτή την ειρηνευτική διαδικασία, σε αυτή την πορεία μας προς την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και την δημοκρατία. Αφιερώνουμε αυτό το βραβείο σε όλες τις επιζήσασες από εγκλήματα σεξουαλικής βίας στο Καγκό αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Είμαστε πεπισμένη ότι η αλλαγή θα έρθει από αυτές τις γυναίκες, τις θαραλέες, τις αποφασισμένες, τις αξιοπρεπείς που μας εμπνέουν καθημερινά. Αφιερώνουμε αυτό το βραβείο σε όλους τους υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αγωνίζονται κάθε μέρα και σε πολύ δύσκολες συνθήκες και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας για να ενθαρρύνουν ένα πνεύμα ειρήνης, την κουλτούρα της ειρήνης, να βοηθήσουν τα θύματα να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Θα ήθελα να χαιρετήσω τον επαγγελματισμό και την αφιέρωση του προσωπικού του πάντσι... καθώς και ε, τον επαγγελματισμό και την ε, προσωπική αφιέρωση στη δουλειά τους ε, όλων των εταίρων μας που μας έχουν βοηθήσει να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Και μάλιστα αναφέρομαι εδώ κυρίως στην ανθρωπιστική υπηρεσία ΕΚΟ, η οποία μας στηρίζει εδώ και 10 χρόνια. Χωρίς εσάς δεν θα είχαμε φτάσει μέχρι εδώ σήμερα. Μαζί, οι ηθήνοντες για τις πολιτικές αποφάσεις, η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών, οι πολίτες, οι άνδρες, οι γυναίκες, όλοι μαζί πρέπει να χαράξουμε μια κόκκινη γραμμή σε σχέση με την προσφυγή στο βιασμό ως όπλος που χρησιμοποιείται στο πόλεμο, προκειμένου να χτίσουμε ένα καλύτερο μέλλον, προκειμένου να μπορέσουμε να προσφέρουμε στα παιδιά και στα εγγόνια μας ένα ασφαλές πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορέσουν να αναπτυχθούν. Έτσι ώστε επίσης να επιτρέψουμε σε όλους αυτούς που έχουν υποφέρει να ατενίσουν το μέλλον με μεγαλύτερη ε, φιλοδοξία. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί ευρωβουλευτέ, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω κάπου εδώ ε, απευθύνοντας το λόγο στους πολίτες της δικής μου χώρας. Αγαπητοί συμπατριώτες, το έθνος μας, η λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό μας ανήκει. Η φυσική και ανθρώπινη πόρη της χώρας μας, τα θεσμικά της όργανα, η μοίρα της, το προμένο της, είναι πράγματα που ε, έχουν να κάνουν με τη δική μας προσωπική ευθύνη. Εμείς οι ίδιοι, ο λαός του Κονγκό πρέπει να... Ε, πρέπει να διατυπώσουμε τους νόμους μας, πρέπει να θεσπίσουμε πλαίσιο δικαιοσύνης και σωστής διακυβέρνησης, το οποίο θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα όλων και όχι μόνο ορισμένων. Το βραβείο Ζαχάροφ που λαμβάνουμε από πλευρά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανήκει στο λαό του Κονγκό, ανήκει σε εσά. Είναι το σύμβολο τη ελευθερία του σκέπτεστε. Είναι ένα δικαίωμα που μα έχει αφαιρεθεί. Είναι ένα δικαίωμα το οποίο ε, μετά από την τρομοκρατία και την καταπίεση που έχουμε βιώσει φαίνεται ενίοτε να έχουμε παρετηθεί από αυτό το δικαίωμα δυστυχώς. Είναι όμως ένα κεκτημένο δικαίωμα και μέσω των εκλεγμένων αντιπροσώπων τους οι λαοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας απονέμουν σήμερα αυτό το βραβείο τίνοντάς μας το χέρι έτσι ώστε να μας βοηθήσουν. Θέλουν να μας στηρίξουν στον αγώνα που κάνουμε εμείς οι πολίτες του Κονγκό για ελευθερία, για ειρήνη, για δικαιοσύνη, για πρόοδο. Σήμερα λοιπόν και ενώπιον ολόκληρου του κόσμου η Ευρώπη μας εκφράζει την αλληλεγγύη ε, της. Η Ευρώπη θέλει να συμβαδίσει, να προχωρήσει μαζί μας σε αυτή την αναζήτηση ε, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στη χώρα μας. Ας ενωθούμε, ας περπατήσουμε, ας προχωρήσουμε προς την Ευρώπη έτσι ώστε η ειρήνη και η δικαιοσύνη, να αποκατασταθούν στο Κονγκό, να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον. Η χώρα μας είναι ένας ασθενής, όμως μαζί όλοι εμείς οι πολίτες και μαζί με τους φίλους μας στον υπόλοιπο κόσμο μπορούμε ε, να τη θεραπεύσουμε. Και θα το κάνουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ.